συνόδου που διακόπη στις 27 Φεβρουαρίου. Τα πρακτικά της ω στις 27 Φεβρουαρίου είναι στη διαθέσή σας. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι. Κυρίες και κύριοι, η Ραζάμ Ζάιτσουνου ε, τιμηθήσαμε το βραβείο Ζαχάροφ πριν από δύο μήνες